Καλησπέρα σα. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι ερωτήσει προ την Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να σα καλωσορίσω. Ξεκινάμε τον κύριο Παπαστάμκο. Έχει την πρώτη ερώτηση, η οποία απευθύνεται ε, στην ε, Επίτροπο για την ανθρωπιστική βοήθεια που πάει στην Βόρεια Αφρική. Thank you, Madam President. Uh, the uh, 3 εκατομμύρια ευρώ επίγουσα βοήθεια για, τις, για τη Λίβη. Χρησιμοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν άμεσα τα ποσά αυτά και μάλιστα ήταν το πρώτο μεγάλο ποσό που έφτασε. Αυξήθηκε στα 30 εκατομμύρια ευρώ στις 3 Μαρτίου λόγω των ανθρωπιστικών αναγκών που διαπιστώθηκαν και έχουμε ένα επιπλέον ποσό 6 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο επίσης έχει κινητοποιηθεί υπό τη γραμμή του προϋπολογισμού για την προστασία των αμάχων και αυτά μαζί με όσα έχουν προσφέρει τα κράτη-μέλη. Η ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διοχετεύεται μέσω της ΕΚΟ ή μέσω της εισίδος βοήθειας που προσφέρουν τα κράτη-μέλη ή μέσω του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βοήθεια λοιπόν σε όσους φεύγουν από την Λιβύη και βρίσκονται στα σύνορα με την Ισία Αλγερία και Αίγυπτο, επαναπατρισμός πολιτών ε, τρίτων χωρών προς την χώρα καταγωγής, προστασία σε όσους έχουν το καθεστώς πρόσφυγα που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους και προς τους πολίτες της Λιβύης που εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Επίσης, ε, έκτακτη βοήθεια από τα αποθέματά μας για την Λιβύη, ιατρικό υλικό, επισητιστική βοήθεια. Και αυτό βέβαια θα χορηγηθεί όταν ε, όλη η χώρα είναι ανοιχτή σε εμάς, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόσβαση σε όλες τις περιοχές. Εν τω μεταξύ, εμείς ε, μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε στο δυτικό τμήμα, αλλά εκεί που βρίσκονται τα στρατεύματα του Καντάφη δεν έχουμε πρόσβαση. Το Μάρτιο έχουμε την ανακοίνωση από την ΑΦΕΤ για την ευημερία στην Νότια Μεσόγειο, όπου έχει μια στρατηγική για την Ευρώπη, έτσι ώστε να στηρίξουμε τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται στις χώρες στην ε, λεκάνη της Μεσογείου. Θέλουμε να στηρίξουμε και την Ιταλία και άλλα κρατημέλη στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσουν τεράστια κύματα μεταναστών από τη Βόρειο Αφρική. Επαναλαμβάνω στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί πως υπάρχουν τέτοια κύματα. Οικονομική βοήθεια και μέτρα, η Frontex, τις κοινέ ε, επιχειρήσει το Χέρμες ε, του 2011 που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο κάλεσε εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη να συμμετάχουν και αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε ε, και προετοιμαζόμαστε για τις διάφορες εναλλακτικές υποθέσεις που ενδέχεται θα παρουσιαστούν έτσι ώστε να καλύψουμε μια πιθανή γκάμα εξελίξεων. Χρησιμοποιούμε πόρους από το Ταμείο για παράδειγμα εξωτερικών συνόρων όπως επίσης και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών είναι έτοιμα να στείλουν ε, προσωπικό και ιατρικό υλικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή οι τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν επηρεάσει ε, την ανθρωπιστική πρόσβαση γιατί όπως σας είπα από την αρχή της κρίσης ε, είμαστε περιορισμένοι στις περιοχές που δεν ελέγχονται από τον Καντάφη και οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρχών ε, στην Τρίπολη και στον Οργανισμό Ηνωμένων Αθνών δεν έχουν δώσει συμφωνία για ανθρωπιστική τουλάχιστον πρόσβαση στις δυτικές περιοχές της Λιβύης. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κύριε Παπαστάμκο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για την εμπεριστατωμένη απάντησή της. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, ότι δείχνει το ανθρωπιστικό της ε, πρόσωπο. Υπάρχει ένα ερώτημα βεβαίως κατά πόσο διαχρονικό είναι το ερώτημα κατά πόσο η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει ε, στα χέρια των πραγματικών ε, αποδεκτών ε, και η διαφάνεια εν προκειμένου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. συγκρατώ κυρία επίτροπε την ευαισθησία βορειοευρωπαϊκών χωρών για να ανοίξει πέρα από το συμβατικό πλαίσιο η ευρωπαϊκή αγορά τα σύνορά της στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από αυτές τις χώρες της Βορειοαφρική στην ευρωπαϊκή ένωση. όμω δεν μπορεί ο ευρωπαϊκό νότο γιατί εκεί με εντοπίζεται ο ανταγωνισμό να πληρώσει για μία ακόμη ε, φορά. δέχεται τι μεταναστευτικέ πιέσει δεν μπορεί να έχουμε πρόβλημα και στον ευρωπαϊκό αγροτικό νότο. σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαστάμκο, γνωρίζουμε όλους τους κανόνες, είναι 32 δεύτερα κανονικά συμπληρωματική. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας από την αρχή, μόλις ξεκίνησε η κρίση. οι πιο δραματικές ανθρωπιστικές επιπτώσεις ε, αφορούν τρία σημεία. Πρώτον, η μεγάλη έξοδος των ε, μεταναστών εργαζομένων ε, προς τον Ήγυρα και προς την ε, Αίγυπτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω κατά αυτή την έννοια υπήρξε αποτελεσματική. Κινητοποιήσαμε ένα εναέρια και θαλάσσια μέσα που προσέφεραν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να επαναπατρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς και επίσης ε, είχαμε ε, και βοήθεια ε, ανθρωπιστική βοηθώντας δηλαδή συγκεκριμένα την υποτιαρμοστία των, για τους πρόσφυγες και πρέπει να πούμε ότι είχαμε πάνω από 20.000 ανθρώπους που φύγανε άμεσα από την Λιβύη. Επίσης στην Ανατολική Λιβύη στην οποία έχουμε πρόσβαση δώσαμε ιατρική βοήθεια ε, καθώς επίσης ε, και ε, δημιουργήσαμε κέντρα διανομής της επισητιστικής βοήθειας. Περίπου 90% της επισητιστικής βοήθειας προέρχεται από εμά. Επίσης, βοηθούμε τους πολίτες της υποσαχάριας Αφρικής, κυρίως τους πολίτες του Τσάντ που βρεθήκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω ε, της ε, ιδιαίτερης επικινδυνότητας. Δηλαδή υπήρχε η υποψία ότι ήταν μισθοφόροι και επομένως έπρεπε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε ε, να τους επαναπατρίσουμε ασφαλώς κυρίως στην περίπτωση της Αιγύπτου. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι σαφώς υπάρχουν πολλές ανθρωπιστικές ανάγκες στις περιοχές τις οποίες ελέγχει ο, ο Καντάφη. Έχουμε ήδη ε, δημιουργήσει ένα απόθεμα 9 εκατομμυρίων ευρώ έτσι ώστε οποτεδήποτε μπορέσουμε, οποτεδήποτε έχουμε δυνατότητα πρόσβασης να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, αυτό είναι ακριβώς η, ε, το, το κέντρο της ε, ε, πολιτικής μας για αυτό το κομμάτι της Μεσογείου. Βεβαίως είναι ακριβώς η βάση για την δημιουργία μέλλοντος για τις χώρες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δίνουμε μεγάλη έμφαση στο εμπόριο. Εμπόριο βεβαίως με την Ευρώπη αλλά και μεταξύ των άλλων χωρών της Μεσογείου. Ευχαριστώ. Έχω και άλλη συμπροματική του κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, όντως η παρούσα κατάσταση στις χώρες της Βορειοαφρικής σημαίνει μεγάλες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοσιεύτηκαν άθρα στους Financial ε, Times που λέγουν ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επαναπατρίσει τους δικούς τους πολίτες, αλλά έχουν αφήσει εκεί κόσμο ε, και πολλούς ε, Βουλγάρους ε, χωρίς καμία... Μάλλον επειδή έφυγαν οι Βούλγαροι που ήταν νοσηλευτικό προσωπικό, έχει μείνει ο κόσμος εκεί χωρίς περίθαλψη. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε. Okay. Um, Επιτρέψτε μου να σας πω καταρχάς ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επαναπατρίστηκαν με μεγάλη επιτυχία, συντονίστηκαν για την εκένωση τα κράτη-μέλη και είχαμε ένα ε, κέντρο ελέγχου και πληροφόρηση για το συντονισμό αυτό. Ως αποτέλεσμα, ε, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών μας ε, βγήκε από τη Λιβύη με τον πιο ασφαλή και ταχύ τρόπο μέχρι που ολοκληρώθηκε η μαζική εκένωση, μόλις 200 ε, παρέμειναν 200 από εκείνους που, ήθελαν να φύγουν και στο μεταξύ ε, με ένα ρωσικό αεροπλάνο έχουν φύγει περισσότεροι. Το θέμα του ιατρικού προσωπικού και της περίθαλψης βεβαίως ε, μετά την εκένωση των Ευρωπαίων πολιτών είχαμε και συνέπειες, διότι ορισμένοι ε, από τους Ευρωπαίους πολίτες ήταν νοσηλευτικό προσωπικό και ήταν ε, μέλη εργαζόμενοι στο Λιβικό Σύστημα Υγείας. Ιδιαίτερα νοσηλεύτριες, όχι τόσο πολλοί γιατροί, νοσηλεύτριες. Και εκεί ακριβώς ε, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αυτή τη στιγμή έτσι ώστε οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που ασχολούνται με την ιατρική περίθαλψη να παρέχουν αυτή την υπηρεσία σε ε, Λιβύους πολίτες στη Λιβύη. Για μας ε, ε, τονίζουμε πολύ το θέμα της πρόσβασης στη Δυτική Λιβύη. Δυστυχώς ο Καντάφη δεν αφήνει στη Δυτική Λιβύη το προσωπικό αυτό να Στείλαμε πυρογνώμονες για μια ερευνητική αποστολή εξεταστική των πραγμάτων και μας είπαν ότι υπάρχουν και τραυματίες που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Ε, υπάρχει και προσωπικό, υπάρχει και εξοπλισμός ιατροφαρμακευτικός επαρκής ε, στην Ανατολική Λιβύη μεν. Πλην όμως στη Δυτική Λιβύη, ε, στη Μισράτα και δυτικά της Μισράτα που είναι υπό τον έλεγχο του Καντάφη δεν επιτρέπει την είσοδο. Και όπως μπορείτε να γνωρίζετε φαντάζομαι γίνονται απόπειρες τώρα ε, δια θαλάσσης να έχουμε πλωτά ε, νοσοκομεία ε, για να βοηθήσουν στην ιατροφαρμακευτική περιθέψη. Ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση, αυτή του κυρίου Μπαλτσίτης, προς την κυρία Δαμανάκη. Λοιπόν, σας δίνουμε ένα λεπτό για να αλλάξετε θέση. Έχουμε εδώ πέρα μια ερώτηση λοιπόν σχετική με τις ανισότητες στα κράτη-μέλη όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Κύριε Επίτροπε, όταν είστε έτοιμοι μπορείτε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα όσα έχουμε στη συνθήκη, η αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ε, δρομολογεί δράσεις για να στηρίξει ή να συμπληρώσει τις δράσεις των κρατών μελών για να προστατεύσουν και να βελτιώσουν την ανθρώπινη υγεία. Του δουλεχθέντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει πως όλοι οι πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχουν καθολική πρόσβαση σε ε, υπηρεσίες περίθαλψης υψηλής ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει ξεκινήσει αρκετές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Θα απαντήσω λοιπόν σε οτιδήποτε με ρωτήσει επιπλέον ο Ευρωβουλευτής. Το 2009 έχουμε την ανακοίνωση για την αλληλεγγύη στην υγεία, μείωση των ε, ανισοτήτων στον κλάδο της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση αυτή τονίζει την ανάγκη που υπάρχει να γεφυρώσουμε τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Πέρσι το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των υπηρεσιών της ξεκίνησαν μια κοινή δράση με 14 κράτη-μέλη για να μειωθούν οι ανισότητες στον κλάδο της υγείας στα πλαίσια του προγράμματος υγείας που τρέχει. Η καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην υγεία αποτελούν και το στόχο της συντονισμού που γίνεται για την υγεία μακροπρόθεσμα και στο πλαίσιο αυτό τα κράτη-μέλη συμφώνησαν συγκεκριμένους στόχους για τα συστήματα περίθαλψης. Η πρόσβαση στην περίθαλψη, η ποιότητα αυτής της περίθαλψης και επίσης η βιωσιμότητα ε, των πολιτικών. Επιπλέον, μέσω της νέας οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών ε, στην διασυνοριακή προσφορά υπηρεσιών περίθαλψης δίδεται η δυνατότητα ε, να πληροφορηθεί κανείς ε, τι είδους θεραπείες είναι διαθέσιμες στο εξωτερικό και δίνεται να ζητηθεί και η αποζημίωση της δαπάνης σε περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες. Στην πολιτική συνοχή έχουμε κάποια μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται και είναι ο εξυγχρονισμός της υποδομής της νοσοκομιακής, αγορά ιατρικού υλικού και εξοπλισμού και εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν να ε, βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών ε, στις υπηρεσίες περίθαλψης και κυρίως στις φτωχότερες περιοχές. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ ο κ. Μπαλτσίτης. E, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, είμαι ευγνώμων για την συνολική σας απάντηση, όμως οι ψηφοφόροι μου συχνά με ρωτούν όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν περίπλοκες ασθένειες, το κεντρικό ερώτημα είναι βεβαίως το θέμα ε, της περίθαλψης, ε, αλλά και το τι συμβαίνει με τους συνοδούς τους. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν, περιθάλπτουν ε, αυτούς τους ασθενείς, μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική προστασία και για αυτούς που προσπαθούν έχουν τους ασθενείς. Θέλετε να απαντήσετε, μάλλον όχι, να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις μαζί, λέει η Πρόεδρος. Ο Αντές και μετά Ματέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ε, με δεδομένο ότι η οδηγία στην οποία αναφερθήκατε για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ θα ήθελα να σας ρωτήσω έχει το δικαίωμα από τώρα ο ασθενής στην περίπτωση που αναζητήσει υπηρεσίες υγείας σε άλλο κράτος να αποζημιώνεται από τα ταμεία του. θυμίζω απλώς ότι σχετικές θετικές αποφάσεις έχει πάρει ήδη το ευρωπαϊκό δικαστήριο. ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Εγώ ε, θέλω να κάνω ε, ερώτηση για τους αλλιευτικούς πόρους. Σήκωσα σε λάθος στιγμή το χέρι μου. Ε, εντάξει κυρία Τικάου, τότε ελάτε και θα σας επιτρέψω να θέσετε το ερώτημά σας. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε θα ε, ήθελα να πω ότι δυστυχώς πολλές χώρες μειώνουν τον προϋπολογισμό τους που αφορά τα θέματα υγείας λόγω της κρίσης. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τον προϋπολογισμό ε, υγείας των κρατών μελών γιατί είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επιτροπέ, αυτό που μπορώ να πω σε γενικέ γραμμέ είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μην λησμονούμε ότι εδώ η αρμοδιότητα ε, είναι των κρατών μελών. Θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Και βεβαίω καταλαβαίνω τις, ε, τα επιχείρηματά σα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Παρ' όλα αυτά όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι προβλέπεται, αλλά παρόλα αυτά ε, θα προσπαθήσει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εναρμονιστεί η κατάσταση. Προτεραιότητά μα είναι να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε αυτές, να μειωθούν αυτέ ε, ε, οι διαφορέ. Επίση, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας όσον αφορά την, το, το, την πρωτοβουλία ευθύνη ευθύνη, ε, εταιρική ευθύνης των φαρμακοβιομηχανιών. Ε, στον κύριο Κουντή μπορώ να πω ότι όταν θα εφαρμοστεί η οδηγία τότε ε, θα έχουμε ένα σαφές πλαίσιο ε, σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων που έχουν δοθεί για διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας. Θα δούμε βεβαίως και τι έκβαση θα έχουν οι περιπτώσεις οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης γιατί ε, αυτή τη ε, στιγμή ε, όντως δεν ισχύει η επιστροφή των χρημάτων. Μέχρι τότε θα πρέπει να περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι ερώτηση Χόκκινε και αφορά τον Επίτροπο Ταγιάννη. Σχετικά με τις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε όσον αφορά τις τεχνολογίες ε, γενικής ε, εφαρμογής την 30 ε, Σεπτεμβρίου του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει μια ανακοίνωση η οποία αφορούσε κοινή στρατηγική για τον τομέα αυτό. Στην ανακοίνωση αυτή εμείς ε, ε, καταδεικνύαμε ότι παρά τις εξαίρετες ε, προϋποθέσεις έρευνας και ανάπτυξης βασικών τέτοιων τεχνολογιών, δυστυχώς δεν καταφέρνουμε να έχουμε την ανάλογη επιτυχία όταν δηλαδή τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικές υπηρεσίες ή συγκεκριμένα αντικείμενα, προϊόντα. Επομένως, πρέπει να ακολουθήσουμε στρατηγική ε, η βάση των οποίων οι τεχνολογίες γενικής εφαρμογή να βρίσκουν πραγματική εφαρμογή στην ε, βιομηχανία. Αυτό έχει υπογραμμιστεί και στις ε, κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την καινοτομία και την ψηφιακή Ευρώπη. Στην ανακοίνωση Επιτροπής του Ιουλίου 2011 δημιουργήθηκε, βάσει αυτής της ανακοίνωσης, δηλαδή δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Επικυρώθηκε η ομάδα αυτή από τρεις επιτρόπους, την κυρία Νέλη Κρούς, την ε, κυρία Μάρια Κουίν, ε, καθώς επίσης και τον υποφαινόμενο η ομάδα αυτή έχει εντολή ενός έτους έτσι ώστε να υποβάλει συστάσεις για τα πολιτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν έτσι ώστε οι τεχνολογίες γενικής εφαρμογής ε, να ε, μπορέσουν να προωθηθούν στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια ομάδα που, που απαρτίζεται μάλλον από εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, από εκπροσώπους των τεχνολογικών γενικής εφαρμογής, από εκπροσώπους γενικής ε, και ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τον Φεβρουάριο αυτή η Επιτροπή υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα προσχέδιο το οποίο αναφέρει τα κύριε, τις κύριες προκλήσεις ε, το, της μετάβασης των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής σε προϊόντα το site της Γενικής Διεύθυνσης ε, Επιχειρηματικότητας μπορεί κανείς ε, ε, να βρει το κείμενο αυτό. Και τον Ιούλιο του 2011 θα υποβληθεί η τελική έκθεση της ε, ομάδας ε, αυτής ε, που θα αποτελέσει βεβαίως βάση σκέψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα αποτελέσει λοιπόν μια βάση για την προώθηση των τεχνολογιών και της καινοτομίας. Αυτές οι τεχνολογίες βεβαίως και πρέπει να το αναγνωρίσουμε είναι της σημασία για την οικονομία μας και μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την δημιουργία νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών και που θα μπορέσουν να αποτελέσουν την νέα βιομηχανική μας βάση, αυτό που θα, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε νέα βιομηχανική επανάσταση. Ε, με τον τρόπο αυτό η βιομηχανία μας θα γίνει πιο ανταγωνιστική και θα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος ε, μιας ε, οικονομίας που θα κάνει λογισμένη χρήση των των μορφών ενέργειας, αποτελεσματική χρήση όλων των καινοτομιών και ε, περιβάλλον που δεν θα χρησιμοποιεί δημοξίδιο του άνθρακος. Διαφορετικά θα χάσουμε, αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες, θα χάσουμε πολύ. Αυτές οι τεχνολογίες αποτελούν βάση για το μέλλον και την ανάπτυξη. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με τις ε, εκτιμήσεις μας, ο όγκος τους Ε, κυμαίνεται από 950 μέχρι 1 δις 100 εκατομμύρια. Και ε, η βάση τους μπορεί να φτάσει μέχρι το, η χρήση τους μπορεί να, να, φτάσει μέχρι το 46% ε, των νέων τεχνολογιών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ε, ρόλο και να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στην βιομηχανία και επομένως πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο δεν μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να παίξει σωστά τον ρόλο της. Χρειαζόμαστε βεβαίως την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολύ περισσότερο μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, όπου έδωσε ε, περισσότερες ε, δικαιοδοσίες στο Κοινοβούλιο. Και εγώ σαν παλαιός Ευρωπαίος βουλευτής λέγω ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου οπωσδήποτε θα μας οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα και σε αυτόν τον τόσο θεμελιώδη για την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή οικονομία τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χάρκιν, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας και συγχαρητήρια ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο σας που προσπαθείτε να παραμείνετε εχμή του δόρατος της ε, νέας ε, βιομηχανικής επανάστασης. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει η λεγόμενη κοιλάδα του θανάτου που ε, χωρίζει την εφεύρεση από την εφαρμογή της και την κυκλοφορία στην αγορά. Και επίσης ε, υπάρχουν προβλήματα ε, όπως είναι το ε, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Τεχνίας για τα θέματα της πληροφορικής και το ανάλογο κανονιστικό πλαίσιο. Τι βήματα έχει κάνει, αν έχει κάνει τέτοια βήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει κάποιο από αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρκιν γιατί υπογραμμίσατε και την εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά βεβαίως ζητάτε ταυτόχρονα και μεγαλύτερη δέσμευση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ε, σε αυτήν την φάση εμείς περιμένουμε ε, τις προτάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων που ανέφερα και προηγουμένως ε, πριν προωθήσουμε ολοκληρωμένη στρατηγική ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ενδιάμεσο έγγραφο εργασίας η ομάδα των εμπειρογνωμόνων πρότεινε τρεις πυλώνες έτσι ώστε να καλυφθεί ε, αυτή η απόκληση της ε, καινοτομίας ε, και βεβαίως μονάχα εάν αυτές οι τεχνολογίες μπορέσουν να εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη θα είμαστε ικανοποιημένοι υπάρχουν πρωτότυπα όντως τα οποία καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, και θα πρέπει να είναι στοχευμένα στην τεχνολογική έρευνα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ε, δημιουργία προϊόντων. Βεβαίως οι εφευρέσεις ε, και οι τεχνολογικές κατακτήσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε ανταγωνιστικά προϊόντα και επομένως χρειάζεται εξισορρόπηση μέσω προγραμμάτων επίδειξης και προϊόντων επίδειξης ε, τρίτον, η Ευρώπη θα πρέπει να διατηρήσει τις ε, παραγωγές της δυνατότητες αλλά να δημιουργήσει και νέες τέτοιες ικανότητες έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική και όσον αφορά τις δάσεις και όσον αφορά τις τιμές ε, και να δημιουργηθεί ένα σωστό πλαίσιο για τους επενδυτές έτσι ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά κοινοτικά προγράμματα τα οποία ευνοούν και μπορούν περαιτέρω να ευνοήσουν ρυθμίσουν αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να καλύψουμε ε, το κενό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην έρευνα και την εφαρμογή ε, και που είναι χαρακτηριστική και πολλών άλλων ε, τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πέρασμα λοιπόν από την έρευνα στην εφαρμογή είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλο το βιομηχανικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς εγώ είμαι υπέρ και άλλωστε έχουμε ε, έχουμε στηρίξει την πολιτική των κλάστερς ε, πρέπει να πούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 2.000 ε, κλάστερς αυτή τη στιγμή γιατί θέλουμε να διασυνδέσουμε σωστά την έρευνα, την καινοτομία και την βιομηχανία για να μπορέσουμε από την έρευνα να περάσουμε στην βιομηχανική εφαρμογή. Ε, σας διαβεβαιώ κυρία Χάρκιν ότι θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε, ε, θα εξακολουθήσουμε να μελετούμε όλες τις προτάσεις που μας υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ προσωπικά τις μελετώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίω θα αποθυσαυρίσω όλες αυτές τις προτάσεις που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ Επίτροπε. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη ερώτηση του κυρίου Ντέιβις και απευθύνεται στην κυρία Δαμανάκη. Και αυτή τη φορά πρόκειται για το μέλλον της αλληλευτικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, κυρία Πίτροπε. Okay, thank you. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν οι υπηρεσίες μου άρχισαν να ε, ετοιμάζουν τη δέσμη μέτρο για τη μεταρρυθμίση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ε, προέβησαν σε μια βαθύτατη αξιολόγηση διαφόρων δυνατοτήτων. Η μία ε, δυνατότητα που είχαμε και επιλογή είναι να συνεχιστεί η παρούσα πολιτική και μετά το 2013. Αυτό το status ε, quo χρησιμοποιήθηκε ως ε, ορόσημο για τη συγκριτική αξιολόγηση, benchmark λοιπόν, για να εκτιμηθούν και οι υπόλοιπες δυνατότητες με μακροπρόθεσμα ε, μέτρα, σχέδια ελέγχου και ε, διαχείριση ε, της λαθραλίας ή της μη δηλωμένης αλίας. Είναι σαφής η κατάσταση πάντως, εάν δεν αλλάξουμε πολιτική, μέχρι το 2020 η αηφορία των αλευτικών αποθεμάτων γενικά αποκλείεται. Και σε ό,τι αφορά ε, την αηφορία και τη βιωσιμότητα από πλευράς περιβάλλοντος, μόλις το 6% των αποθεμάτων που μελετήθηκαν μέχρι το 2020 θα έχουν φτάσει σε επίπεδα ανανέωσης και ε, αηφορίας. Έχουμε δε και την υποχρέωση μέχρι το 2015 να εξασφαλίσουμε την πλήρη βιωσιμότητα. Επαναλαμβάνω, ε, συνεχίσουμε την κατάσταση που ισχύει σήμερα, σε καμία περίπτωση δεν θα φτάσουμε το στόχο του 2015 για την ανανέωση των ε, ειδών. Σε ό,τι αφορά την οικονομική επίδοση τώρα των αλληλευτικών μας στόλων, υπό το σενάριο του status quo μόνος ε, ορισμένα, σκάφη ορισμένη στόλη ε, θα το πετύχουν αυτό το στόχο, ενώ κάποιοι άλλοι ε, θα έχουν μηδενικό αποτέλεσμα. Για την κοινωνική βιωσιμότητα είναι η ίδια εικόνα. Θα μειώνεται ε, η απασχόληση στον τομέα της αλίευσης, οι μισθοί θα παραμένουν χαμηλοί και το επάγγελμα του αλία θα είναι όλο και περισσότερο ε, εχθρικό και καθόλου ελκυστικό για τους ε, νέους. Για μας λοιπόν η συνέχιση της παρούσης κατάστασης δεν είναι για μας επιλογή. Χρειαζόμαστε τη μεταρρύθμιση και θα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Ντέιβις και άλλες δύο συμπροματικές θα τις ομαδοποιήσουμε για να απαντήσει στη συνέχεια συνολικά η Επίτροπος. Ο κύριος Ντέιβις. Η Επίτροπος λοιπόν μας περιέγραψε μια εξαιρετικά απογοητευτική κατάσταση γιατί αν δεν κάνουμε τίποτα τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης για τους αλληλείς και ο κλάδος θα μαραθεί. Όμως μπορεί να έχουμε κάποια εναλλακτική λύση η οποία θα είναι καλύτερη γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με το 50% της αλληλευτικής ε, προσπάθειας. Τα αποθέματα είναι χαμηλά γιατί είχαμε υπεραλλήλευση για δεκαετίες. Η πραγματικότητα είναι η εξής η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι. Κύριε Επίτροπε, εσείς δεν μπορείτε καν να αποκλείσετε τη δυνατότητα, εάν συνεχίσουμε έτσι όσο έχουμε, αρκετά από αυτά τα αποθέματα να εξαφανιστούν. Έχουμε από την κυρία Ματέρα και από τον κύριο Κέλλη κάποια αιτήματα για να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου ξαναδώσετε το λόγο. Σημερίζομαι ε, την ανησυχία των ε, συναδέλφων για, τις για τους πόρους ε, στην Μεσόγειο και την διατηρήση των οικοσυστημάτων στην Μεσόγειο. Αλλά βεβαίως οι κοινωνικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν τα, μπορεί να έχει παρούσα κατάσταση ε, κυρίως ε, δε σε ορισμένες ε, κοινωνίες οι οποίες εξαρτώνται από την αλία θα πρέπει να μας οδηγήσει στην προστασία αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν μόνο με τη θάλασσα. Ευχαριστώ είναι πραγματικά απογοητευτική η κατάσταση που μας περιγράφεται και ένα από τα προβλήματα που αναφέρει ο κύριος Ντέιβις ε, στην ερώτηση είναι το θέμα των απορρίψεων. Πρόσφατα συναντήθηκα με ένα αλλιέα και μου είπε ότι έχει βρει ε, ένα νέο δίχτυ, έχει εφεύρει ένα νέο δίχτυ για την αλία του τόνου που μειώνει τις ε, απορρίψεις. Αυτό πώς το αξιολογείτε εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κυρία Πίτροπος. Εάν συνεχίσουμε ε, όπως κάνουμε σήμερα, ναι, έχετε δίκιο. Αντιμετωπίζουμε τη δυνατότητα της ε, εξαφάνισης πολλών ειδών, πολλών αποθεμάτων, αναμφίβολα. Και θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι πολύ ευαίσθητη η κατάσταση. Εάν λοιπόν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, ξέρετε πως οι συνέπειες θα είναι ενδεχομένως εξαιρετικά κακές. Γι' αυτό χρειάζεται η μεταρρύθμιση και για το λόγο αυτό θα εξετάσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε μια πραγματική ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας αποθεμάτων και βέβαια κοινωνικο-οικονομικής ε, και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που θα έχει μεταρρύθμιση. Αλλά θέλω να σας ξεκαθαρίσω το εξή. δεν έχει να κάνει με δική μας προτίμηση. Δεν είναι ότι εμείς προτιμάμε να φροντίζουμε το περιβάλλον και δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το να φροντίζουμε τους αλλοίς. Όχι. Μας ανησυχεί η τύχη τους και μας ανησυχεί η τύχη των επόμενων γενεών των αλλιέων και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, να είμαι ειλικρινής. Εάν δεν έχουμε αποθέματα να αλλιεύουμε, εάν δεν υπάρχουν πια ψάρια στη Μεσόγειο, και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ύδατα, δεν έχει μέλλον αυτός ο κλάδος. Για να είμαστε λοιπόν σίγουροι πως η αλληλής και η δική μας αλληλευτική βιομηχανία έχει μέλλον, χρειάζεται να κάνουμε μεταρρύθμιση. Αυτό είναι σίγουρο. Πρόκειται λοιπόν να παρουσιάσουμε κάποιες θετικές προτάσεις και θα εξασφαλίσουμε, θα εξασφαλίσουμε στο μέλλον την επαγγελματική ζωή των αλλιέων μας. Τώρα, για την επιλογή των ελευτικών εργαλείων, κάτι το οποίο ανέφερε κάποιος από εσά, να σας πω, είμαστε στη διάθεσή σας και θα εξετάσουμε οποιοδήποτε νέο εργαλείο, οποιαδήποτε καινοτομία ε, για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και στα πλαίσια του νέου συστήματος χρηματοδότησης θα διαθέσουμε πόρους με να το πω έτσι, γενναιόδρο τρόπο παρόλο την κρίση, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι πως τα εργαλεία αυτά θα χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο. Χαιρετίζω λοιπόν όλες τις πρωτοβουλίες από τον κλάδο της ε, αλληλευτικής βιομηχανίας και από τους αλληλείς μας, έτσι ώστε να γίνουν ε, βελτιώσεις ε, σε επίπεδο εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Θα ήθελα να επαναλάβω εδώ πως η τρέχουσα κατάσταση δεν αποτελεί εναλλακτική λύση πλέον. Γιατί? γιατί δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων, γιατί δεν εξασφαλίζει το βίο των αλλιέων μας και των κοινοτήτων των παράκτιων της Ευρώπης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον κύριο Χίγγινς και έχει να κάνει με την απαγόρευση που προτείνεται για τα πτερήγια καρχαρία και την αφαίρεση από το αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο βουλευτή για την ερώτησή του, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ε, για την κοπή των ε, πτέρυγιων του Καρχαρία. Από το 2003 έχει απαγορευτεί ε, μέσω κανονισμού του Συμβουλίου ε, σε ευρωπαϊκά ε, πλοία που αλλιεύουν παντού ε, στον κόσμο και σε γενικότερα πλοία που αλλιεύουν εντό των χωρικών υδάτων τη ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγορεύεται δηλαδή. Δυστυχώς όμως υπό κάποιους όρου και ε, προϋποθέσεις μπορεί στα σκάφη τα ίδια ε, να αφαιρούνται τα πτερίγια κατά τη διάρκεια ε, της κατεργασίας ε, των καρχαριών που έχουν αλλιευθεί και αυτό είναι το πρόβλημα των τελευταίων ετών. Έχουμε το Φεβρουάριο του 2009 υποβάλει ένα πρόγραμμα δράσης και λάβει διάφορα μέτρα. Ε, συνεργαζόμαστε με περιφερειακούς οργανισμούς στενά για να υπάρχει ε, μια διαχείριση των πιο ευάλωτων ειδών καρχαρία για να ε, εξασφαλιστεί η αηφορία τους, η βιωσιμότητά τους και να μην έχουμε υπερεκμετάλλευση. Ποιο είναι το πρόβλημα. Χρειάζεται δημόσια διαβούλευση και ήδη έχει αρχίσει αυτή μήνες τώρα και το αντίστοιχο κείμενο παρουσιάζει τρεις από τις βασικές επιλογές και δυνατότητες που συζητούν παγκοσμίω οι εμπειρογνώμονες για να βεβαιωθούμε για την πλήρη συμμόρφωση και να βελτιώσουμε ε, τους ελέγχους. Πολύ ενδιαφερόμενοι ε, και το κοινό ε, μας έστειλαν τα σχόλιά τους, ε, εργαζόμενοι στον κλάδο, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, επιστήμονες κτλ. Πρέπει να σας πω ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα της προστασίας των καρχαριών και ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να μελετήσουν με ε, μεγάλη επιμέλεια όλες τις προτάσεις που λάβαμε και συνέχεια θα κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου και σκοπιμότητας που χρειάζεται για να αλλάξει ο κανονισμός. Προτείνω το συντομότερο δυνατό να εγκριθεί ε, νομοθεσία, κανονισμός και πρέπει να σας πω ότι για μένα αποτελεί προτεραιότητα αυτό για να μην χάσουμε περισσότερο χρόνο. Ε, πλέον θα ήθελα να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, λάβει πολλά μέτρα για να εξασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των καρχαριών γενικώ. Πέρα από την αφαίρεση των πτερυγίων. Έχουμε υποβάλει πρόγραμμα δράσης και έκτοτε λάβει μέτρα. Έχουμε απαγορεύσει ε, την αλίευση διαφόρων ειδών ε, καρχαρία ε, σε ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε απαγορεύσει και τα δίκτυα άνω των 200 μέτρων για να προστατεύουμε τους καρχαρίες που ζουν σε μεγάλα βάθη. Πάντα η ποσόστος θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Έγινε πολύ σκληρή διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό. Στο τέλος όμως επιτύχαμε και έχουμε μια πρόταση που εξασφαλίζει για φέτος την εφορία και ελπίζω τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χίγκινς, ο κύριος Κρόλη και ο κύριος Ντέιβις ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Είναι ένα βάρβαρο έθιμο να αφαιρούνται τα πτερίγια του Καρχαρία. Είναι απάνθρωπο τα πετάτε, τους πετάτε μετά στη θάλασσα και πεθαίνουν. Πρέπει να απογορευτεί λοιπόν. Και ενώ η Επίτροπος αναφέρθηκε στον κανονισμό του 2003, να σας πω πως δεν εφαρμόζεται. Και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να έχουμε ένα κανονισμό που θα απαγορεύει τελείως αυτή την αφαίρεση, γιατί με τον τρόπο αυτό θα εξαφανιστεί αυτό το είδος. Έχουμε δει τα στοιχεία. Το 2009 26 με 73 εκατομμύρια καρχαρίες έχασαν τα πτερίγια τους και αυτά μπήκαν στο εμπόριο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να απαγορευτεί η εμπορία αυτών των ειδών και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει εμείς να βρεθούμε στην αιχμή του δόρατος. Ευχαριστώ κύριο Κρόλη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Επίτροπο για την απάντησή της. Παρόλο που το 2003 η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία απαγορεύτηκε έχουμε ε, μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που έχουμε για τα, με τα σκουμπριά. Δηλαδή, έχουμε τι γίνεται ε, στην ε, περιοχή του ΕΟΧ και ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Ξέρετε τι έχουν κάνει και στην Ισλανδία και στη Γρυλανδία και το πώς η δική τους υπεραλίευση επηρεάζει τη δυνατότητα λίευσης που έχουν οι ευρωπαϊκοί ε, στόλοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ε, για το σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε τεράστιες ε, προσπάθειες. Εξαφανίζονται τα λιωτάρια από την Αφρική και οι καρχαρίες από τους ωκεανούς μας. Συγχαρητήρια στην Επίτροπο για αυτά που προσπαθεί να κάνει, αλλά ε, αυτό είναι κάτι που ζητάει η αγορά. Ε, η Ασία έχει τεράστια ζήτηση και πολλά τα λεφτά που μπορεί κανείς να κερδίσει. Και ο μόνος τρόπος να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ελέγχουμε και να περιορίσουμε αυτό που συμβαίνει είναι όταν εκφορτώνονται τα πτερίγια να είναι ενωμένα με ε, το σώμα του Καρχαρία. Η Επίτροπος παρακαλώ. I can θα συμφωνήσω με τα μέλη του Συμβουλίου ότι ε, παρότι υπάρχει απαγόρευση ε, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση. Συμφωνούμε γιατί, μαζί σας ε, γιατί η πραγματικότητα διαφέρει. Γνωρίζουμε ότι η βιομηχανία των, της εμπορίας πτερυγίων Καρχαρία δίνει πάρα πολλά χρήματα. Να σας εξηγήσω λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Το πρόβλημα προκύπτει διότι η βιομηχανία τώρα μπορεί ε, να ε, δώσει μπορεί να εκφορτώσει ξεχωριστά και σε διαφορετικούς λιμένες τα πτερίγια και τον ίδιο τον Καρχαρία. Ε, Βεβαίω υπάρχει μεγάλη ζήτηση, κυρίως στην Ασία, για τα πτερήγια και επομένως μπορούν τα πτερήγια να τα εκφορτώσουν σε άλλα λιμάνια ενώ το σώμα του Καρχαρία, το οποίο έχει άλλη ζήτηση, σε διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Θέλουμε ε, να, αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αυτό που μπορώ να σας πω λοιπόν είναι ότι προτιθέμεθα να ε, κάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου ε, μια πολύ φιλόδοξη πρόταση. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε νέο νομικό πλαίσιο όσον αφορά την αφαίρεση και την εμπορία των πτερυγίων ε, καρχαρία έτσι ώστε μία και καλή να τελειώσουμε με την κατάσταση αυτή. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση για το σκουμπρί μπορώ να σας πω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και να υπογραμμίσω ότι ε, τα κράτη-μέλη, τα γειτονικά της περιοχής αυτής ε, ήταν εξαιρετικά ε, διαθέσιμα για συνεργασία και ότι οι αλλοί έκαναν πολλές θυσίες έτσι ώστε να παραταθεί η βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Όμως η Ιρλανδία είχε η, Ισλανδία ε, είχε μια δική της προσέγγιση και μονομερός αύξησε ε, τα ε, ποσοστά της και η Νίση Φερό επίσης. Δεν μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση και ο κύριος Ντεγκούχτ ε, ως αρμόδιος για το εξωτερικό εμπόριο ε, σε συνεργασία με μένα βεβαίως θα υποβάλουμε ε, νέα πρόταση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχει ξεκινήσει διαβούλευση τώρα αλλά τα νομικά εργαλεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην διάθεσή μας αφορά μονάχα το σκουμπρί ε, και όχι τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από το σκουμπρί και αυτά τα προϊόντα ακριβώς είναι ε, τα περισσότερο εξαγόμενα ε, από την Ισλανδία. Επομένως, εμείς θα βελτιώσουμε την κατάσταση ώστε στην επόμενη ελευτική περίοδο να έχουμε την σωστή προστασία των αποθεμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στην ερώτηση του Προέδρου της κυρίας Κράτσα με θέμα τη νέα θαλάσσια στρατηγική της Μεσογείου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. I would like to thank Mrs. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κράτσα για την ερώτησή της, διότι μας δίνει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτή τη τόσο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο. Θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε ανακοίνωση για μια εταιρική σχέση για δημοκρατία και ε, κοινή ευημερία με την νότια όχθη της Μεσογείου. Εκεί αναφέρονται πολλές προτάσεις για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σήμερα γνωρίζει η ε, περιοχή. Είναι η ακραία κατάσταση όπως γνωρίζετε, πολύ ανησυχητική και πολύ εύθραυστη μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Θα ήθελα να πω κυρία Πρόεδρε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη ικανοποίηση ε, παρατηρεί ε, τη γενική αποδοχή της ανακοίνωση αυτής. Με πολύ θετικό τρόπο τη δέχτηκαν όλα τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, ελπίζω. Επιτρέψτε μου τώρα να σας περιγράψω και να σας εξηγήσω κάποιες δράσεις που έχουμε αναλάβει μέχρι τώρα ως προς το στόχο αυτό να έχουμε μια νέα ε, ε, θαλάσσια στρατηγική της Μεσογείου. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ήδη έχουμε στήσει ομάδα εργασίας για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ε, με όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο και τις περιφερειακές οργανώσεις. Και θέλουμε να προχωρήσει αυτό ως εγκάρσια συνεργασία για όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, για τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση επίσης. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ένα πρώτο σχέδιο παραχής τεχνικής βοήθειας το οποίο εντάσσεται στο μέσο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας για την ολοκληρωμένη ε, δράση στη Μεσόγειο. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω το Κοινοβούλιο για μια πρωτοβουλία που ανέλαβα πρόσφατα ένα κοινό πρόγραμμα συνεργασίας στη Μεσόγειο με το ε, Διεθνή Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πραγματικά ποντάρω πάρα πολύ ε, και στις στοχευμένες δράσεις για την ανάπτυξη στη θάλασσα και την ε, κατάρτιση ναυτικών που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Μεσόγειο. Επίσης, θα έχουμε δράσεις που ε, έχουν να κάνουν με ολοκληρωμένη θαλάσσια παρακολούθηση και να συμμετέχει και ο ιδιωτικό τομέας. Γιατί αυτά τα θέματα της θαλάσσης ε, είναι ε, ο θέματα όπου είναι απολύτως απαραίτητη η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτίθεται να υποστηρίξει ένα φόρουμ ακτοφυλακής λιμενικού της Μεσογείου, όλων των χωρών της Μεσογείου και επίσης για τον έλεγχο της αλίας με κατάρτιση εργαστήρια και κοινό έλεγχο σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του ΦΑΟ σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή και σε αυτό το επίπεδο συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, είναι ε, καλό το θαλάσσιο περιβάλλον μέχρι το 2020 σε ανοιχτό επίπεδο και τα κράτη-μέλη συνεργάζονται στα πλαίσια της Σύμβασης της Βαρκελόνης με ε, εταίρους της Μεσογείου για να προλάβουμε τη ρήπανση ε, της Μεσογείου από τα κράτη που βρέχονται από αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ε, προβλήματα της μετανάστευσης και έχουμε εξελίξει την περιοχή, είναι πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει οι γειτονικές μας χώρες που υφίστανται ε, μεταναστευτικές πιέσεις από τον Νότο και μάλιστα με οικονομική υποστήριξη. Ψάχνουμε τώρα επίγουσα βοήθεια ε, από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και δεχομένω και από ένα ταμείο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες καλύτερα ε, για να ε, προσημειώσουμε τα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων συνεργαζόμαστε με τη Frontex και είναι κοινή η προσπάθεια ήδη από το 2011 για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Μαζί με την Europol η Frontex έχει αρχίσει να προετοιμάζει ανάλυση κινδύνου στοχευμένη για να ε, δουν σε ποιο βαθμό η ρευστή πολιτική κατάσταση μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από εγκληματικούς κύκλους. Ευχαριστώ. Η κυρία Κράτσα έχει μια επιπλέον ερώτηση να σα απευθύνει. Και για την αναφορά σα στα, στα σχέδια και τι νέε κατευθύνσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω και για την προσωπική δέσμευση που εκφράσατε και την προετοιμασία σα για αυτή τη νέα πραγματικότητα στη Μεσόγειο. Ήθελα να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα ε, πώ αποτιμάτε τα σχέδια που ήδη έχουν δρομολογηθεί για την απορρίπανση τη Μεσογείου, για τη μεταφορά ενέργεια και πώ αυτά τα εντάσσετε στην ε, σχέση με την θαλάσσια πολιτική. Ε, και τι προστιθεμένη αξία περιμένετε να έχουν τα σχέδια και τα προγράμματα της ε, νέας πολιτικής στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και έχουμε ακόμα μία ερώτηση από τον κύριο Λαβίρ. Δεν ξέρω κύριε Βέγγελ, έχετε κι εσείς ερώτηση σχετική με το θέμα? Yes. Okay. Well, first Mr. Lavia and then Mr. Κύριε Mr. Κύριε Επίτροπε, στα πλαίσια της νέας πολιτικής ε, για τη Μεσόγειο, για την Αλία, στα όσα μας είπατε τώρα για την κατάσταση των χωρών της νότιας όχθης ε, της Μεσογείου που διανύουν μια βαθιά κρίση, η συνεργασία και συγκεκριμένα η διασυνοριακή ε, σε ό,τι αφορά τη συνοχή, χρειάζεται κοινή προσέγγιση γιατί η διασυνοριακή πολιτική και ε, η πολιτική αλίας είναι κάτι που πρέπει να δούμε για να διαφυλάξουμε και τα αποθέματα στη Μεσόγειο αλλά και να ε, επανέλθει η ελευτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η ερώτησή μου σχετίζεται με το γεγονός πως αρκετά κράτη-μέλη προσπάθησαν να μεταφέρουν τα προβλήματα του αλληλευτικού στόλου σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχει. Ε, τουλάχιστον με την νομική έννοια. Μιλάω για την Δυτική Σαχάρα. Έχουμε λοιπόν εντολή αυτή τη στιγμή για την διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Αλίας με το Μαρόκο. Άρα λοιπόν ποιες είναι οι εγγυήσει πως τα χρήματα τα οποία θα λάβουμε βάση τη συμφωνίας αυτής θα ευνοήσουν το λαό της Δυτικής Σαχάρας και δεν θα κανοποιήσει απλώς τις ανάγκες σε αλλιεύμα των Ευρωπαίων αλλιευτών. Θα συμφωνήσω με την κυρία Κράτσα. Η δυνατότητα της ε, ρήπανσης λόγω ενεργειακής μεταφοράς στην Μεσογείο είναι εξαιρετικά υψηλή. Υπάρχει λοιπόν όντως εδώ ένας κίνδυνος. Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και δεν μπορεί να φέρει το βάρος αυτό μιας ενδεχόμενης ρήπανσης. Θα αυξήσουμε λοιπόν και θα βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη ε, και απευθύνουμε προς την κυρία Κράτσα για να της πω πως ο Επίτροπος κ. Ποτότσνικ και εγώ πάμε στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα και θα συζητήσουμε και το θέμα της ρήπανσης Μεσογείου uh, για να δούμε και αυτή τη διάσταση. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλό θα ήταν να μπορούν να ανοιχνεύσουν περισσότερο την ρήπανση από ε, τα καράβια μέσω του EMS και μέσω της ε, ανείχνευσης μέσω δηλοφόρου για το Clean Sinet και το Safe Sinet. Έχουμε αυτά τα δύο συστήματα ε, παρακολούθησης και θα τα χρησιμοποιήσουμε σε όλη τη Μεσόγειο για να δούμε πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ενδεχόμενη ρήπανση που προκαλούν ε, τα διερχόμενα πλοία. Αυτό το λέω γιατί θέλουμε να δώσουμε κίνητρα όχι μόνο στα δικά μας κράτη-μέλη αλλά και στις γειτονικές χώρες μέσω των συζητήσεων που κάνουμε και των συνομιλιών, έτσι ώστε να συνεργαστούμε για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς μέσω της βοήθειας αυτής. Για την περιφερειακή συνεργασία θα απαντήσω το εξή. Ναι, θα αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες και έχουμε μάλιστα αρκετές πρωτοβουλίες στα πλαίσια της Γενικής Επιτροπής Αλληλείας για την περιοχή της Μεσογείου, της GFCM, προσπαθούμε να χαράξουμε μια νέα θαλάσσια στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιωνίου. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις σχέσεις που έχουμε με τα κράτη-μέλη στην περιοχή γύρω από το Ιόνιο και την Αδριατική. Μιλάω για τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Ελλάδα, αλλά επίσης και άλλα κράτη στη γειτονιά, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, συνεργαζόμαστε μαζί τους έτσι ώστε να χαράξουμε μια θαλάσσια στρατηγική που θα βασίζεται στη συνεργασία προ όφελο τη περιοχή αυτή. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω πω αυτό θα αποτελέσει πραγματική ευκαιρία για τα ταμεία συνοχή, όπω μα είπε άλλωστε και το αξιότιμο μέλο του Κοινοβουλίου. Και μία μικρή παρατήρηση για την Δυτική Σαχάρα. Να σα απαντήσω πω όντως έχουμε πάρα πολλέ ανησυχίε που σχετίζονται με το δικαίωμα των πραγματικών δικαιούχων να ευνοηθούν από τα κονδύλια τα οποία εμείς στέλνουμε στο Μαρόκο μέσω αυτής της Συμφωνίας Αλληλείας. Γι' αυτό ζητήσαμε από την μαροκινή κυβέρνηση να μας δώσει στοιχεία που θα αναφέρονται όχι μόνο στην εφαρμογή της συμφωνίας γενικότερα, αλλά και στην περιφερειακή προσέγγιση που ακολουθείται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Επίσης ζητήσαμε να μας εξηγήσουν με ποιο τρόπο γίνεται ο επιμερισμός, η κατανομή μεταξύ περιοχών στο Μαρόκο. Ένα μόνο μπορώ να σας πω πως εμείς θα ανανεώσουμε το πρωτόκολλο για μια μεταβατική περίοδο ενός έτους για να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να το συνεχίσουμε ή όχι. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούμε με ιδιαίτερη σύνεση προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και μπορούμε τώρα να περάσουμε στις ερωτήσεις προς την Επίτροπο κυρία Γκέγγεν Κουίν. Πρώτη είναι του κυρίου Παπα-Νικολάου και αφορά την εκπαίδευση των ερευνητών και αξιολόγηση πανεπιστημίων στην εμβληματική πρωτοβουλία για την καινοτομία. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. on the 3% R&D intensity target. Το 3% του στόχου το ξέρουμε και τα κράτη-μέλη χρειάζονται ε, να ενισχύσουν την ευφυή ανάπτυξη και να αντιμετωπίσουν ε, την πρόκληση. Δείχνει η έρευνα και αξιολόγηση ότι ε, χάνουμε υπολοιπόμεθα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία και η Κίνα τι να μας ξεπεράσουν. Κάλεσε το Συμβούλιο τα κράτη-μέλη να θέσουν ε, φιλόδοξους ε, στόχους για την ε, ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης και να ενισχύσουν τις οικονομίες τους τα κράτη-μέλη πέρυσι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισαν διμερή διάλογο. Τώρα όλα τα κράτη-μέλη έχουν περίπου στόχους εθνικούς ε, για τα σχέδια μεταρρυθμίσεων που θα υποβάλουν μέχρι τέλη Απριλίου του 2011. Στις 12 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση για την ετήσια ανάπτυξη και συμπεριλαμβάνει και τους στόχους για την έρευνα και ανάπτυξη που είναι και ρεαλιστική γενικά και φιλόδοξη και ορίζει ένα νέο κύκλο συντονισμού πολιτικές, ε, εθνικές και ε, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται και ε, αυτό που μας ενδιαφέρει να βγούμε από την κρίση, βέβαια με κάποιους οικονομικούς περιορισμούς ακόμα ζωτικό να φτάσουμε στο στόχο του 3% και αν θέλουμε η Ευρώπη να είναι πιο καινοτόμα θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ε, επιπλέον ε, θέσεις ερευνητών για να φτάσουμε στο στόχο του 3% μέχρι το 2020. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι ερευνητές που χρειαζόμαστε επίσης μέχρι τότε γιατί πολλοί θα βγουν στη σύνταξη και ε, είναι προ όφελο τη κοινωνία και των πανεπιστημίων και τη βιομηχανία. και χρειάζονται ποιοτικά πανεπιστήμια ε, το βαθμολόγιο που χρησιμοποιείται για να συγκρίνει χρησιμοποιεί δείκτες διεθνούς κύρους και τρεις από τους δείκτες αυτοί είναι ε, πόσοι έχουν διδακτορικό από 25 έως 34 ετών σε συγκεκριμένο αριθμό πληθυσμού ε, επιστημονικές ε, δημοσιεύσεις του 10% παγκοσμίω και στο 1 εκατομμύριο πολιτών. Είναι τρεις δείκτες αυτοί, η ποιοτική και ποσοτική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι 37% πάνω από το επίπεδο της Ευρώπης. αύξαν τις επιδόσεις τους. τον Ιούνιο περιμένουμε μια μελέτη σκοπιμότητας για να δούμε μια πολυδιάστατη βαθμολόγηση διεθνή ε, πρόεδρος διακόπτη, δηλαδή πάμε πάρα πολύ. Όχι, δεν σας λέω σταματήστε, απλώς είναι η ταχύτητά σας ηλικιώδης και δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς μας. Πώς θα μπορούσατε να τα πείτε λίγο πιο αργά. Ναι, Πρόεδρε, πάντα τέτοια τα ίδια παθαίνω, λυπάμαι πάρα πολύ. Ε, περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα τον Ιούνιο μιας μελέτης σκοπιμότητας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει μια διεθνή ε, αξιολόγηση ε, πολυδιάστατης και πολυεπίπεδη για να ταξινομηθούν τα ιδρύματά μας και θα καλύπτει επιδόσεις όχι μόνο στην έρευνα αλλά και σε άλλους σημαντικούς τομείς όπως είναι η καινοτομία, η παιδεία, η περιφερειακή ανάπτυξη και η διεθνοποίηση. Πολυδιάστατο ο χαρακτήρας λοιπόν αυτής της έρευνας και θα επιτρέψει σε φοιτητέ ε, ηθήνοντε και τα πανεπιστήμια να επιλέξουν ε, τη διάσταση που θέλουν και ε, τους δείκτες που θέλουν και να κάνουν την ίδια τους προσωπική δαξινόμηση ανάλογα με τις ανάγκες τους. Εκεί συμμετέχουν πάντα όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου παρακαλώ. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Θυμίζω όμως ότι και 8 περίπου χρόνια πριν, το 2003, στο σχεδιασμό μας τότε, στρατηγική για τη Λισαβόνα, λέγαμε περίπου τα ίδια, ότι και τότε έπρεπε να βασιστούμε στην καινοτομία, στην έρευνα και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε και πιο ανταγωνιστική οικονομία. Τι σας κάνει πλέον, είστε πέραν του χρόνου επίτροπο και νομίζω έχετε την εμπειρία να μας απαντήσετε. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά στη νέα στρατηγική που έχουμε για το 2020 θα τα καταφέρουμε και δεν θα έχουμε παρόμοια αποτελέσματα με την προηγούμενη στρατηγική που τελικώ απέτυχε παταγωδός. Συμπληρωματική ερώτηση του κ. Κέλλη. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, είχα κι εγώ ίδιος ε, δυσκολία να παρακολουθήσω την Επίτροπο. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τώρα την Επίτροπο, είναι ικανοποιημένη ε, που έχουν την βούληση και την δυνατότητα ε, και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να ε, συνεργαστούν μεταξύ τους, ε, να κάνουν καλύτερη έρευνα και τελικά να ανεβούν στην ιεράρχηση και την αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Αυτό που διαφέρει τώρα ανάμεσα σε αυτά που δεσμευτήκαμε να κάνουμε βάσει της Λισαβόνας είναι το εξής. Πρώτον, η εκπαίδευση βρίσκεται τώρα στην καρδιά καρδιά, στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής έχουμε δέσμευση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά πλέον και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και επίσης ε, έχουμε 34 δεσμεύσεις όσον αφορά την ε, καινοτομία ε, από ιδιαίτερα κολέγια τα οποία εμείς παρακολουθούμε. Ποιες είναι οι εξελίξεις, είναι, ποιο είναι το τελικό παραχθέν έργο κτλ. Κάθε χρόνο ελπίζουμε ότι θα έχουμε και μία σύμβαση καινοτομία έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί να, να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να ε, συζητήσουν. Ε, η ε, στενότερη εποπτεία που ήταν ακριβώ το ασθενέ σημείο μέχρι τώρα πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα βελτιωθεί. Επίση υπάρχει βάσει των αποτελεσμάτων τη έρευνα η εθνική έρευνα η οποία θα γίνει γίνει σε κάθε χώρα έτσι ώστε ε, να ξέρουμε και από πλευρά των Ιδρυμάτων πώς προτίθενται να επιτύχουν τους στόχους. Εξυγχρονισμός των πανεπιστημίων. Πολύ ευρύ ε, το θέμα και αφορά νομίζω όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας αρκεί να έχουμε ένα-δυο καλά πανεπιστήμια σε κάθε χώρα που βρίσκονται ακριβώς ε, στην κορυφή. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε όλες τις βαθμίδες του πανεπιστημίου και όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και να με επικαλύψεις σαν αυτές που αναφέρατε γιατί κάποια πανεπιστήμια τώρα μπορεί να αισθάνονται ότι είχαν την δυνατότητα αριστείας ε, αλλά όχι σε όλες τις σχολές τους. Ε, Αυτό αυτό όμως δεν είναι δυνατόν εμείς να, δεν είναι δυνατόν εμείς να δεχτούμε μια τέτοια ε, επικάλυψη και έναν τέτοιο κατακαιρματισμό. Ε, αυτό που ε, μπορούμε να κάνουμε και αυτό που κάνει και η Επίτροπος Βασιλείου είναι να εξηγεί στα κράτη-μέλη ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τις στρατηγικές του παρελθόντος. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα δημιουργήσουμε σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια κέντρα αριστείας. Και ε, βεβαίως να εφαρμόσουμε και ένα γενικό ε, πρόγραμμα εξυγχρονισμού των πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση, κύριος Τσουκαλάς. Ελάχιστη έλεγχη και υψηλά ποσοστά λαθών στα έργα του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Επίτροπος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ε, σκεφτώ και τους διερμηνείς. Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των, ε, των οικονομικών ελέγχων είναι να υπάρχει αρκετά μεγάλος ε, αριθμός στοιχείων που δίνουν δικαιούχοι. Για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 2007 με 2013 η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι 18 μήνες μετά την έναρξη του έργου. Ως αποτέλεσμα ε, αριθμός των ε, έργων που μπορούν να ε, ελεγχθούν έφτασε στην κρίσιμη μάζα του το 2010 και μόνο. Στόχος είναι να βεβαιωθούμε για την νομιμότητα και το νομότυπο όλων αυτών των διαδικασιών καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος Πεσίλ. Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε 345 ε, οικονομικούς ελέγχους που ε, καλύπτει πάνω από 400 συμμετέχοντες, 422 περίπου. Οι διορθώσεις οικονομικές φτάνουν, ε, φτάνουν στο 4,48 εκατομμύρια ευρώ από τις συνεισφορές του ε, προγράμματος πλαισίου. Τα προγράμματα αυτά γίνονται με συγχρηματοδότηση, ε, με επιστροφή των ε, επιλέξιμων πραγματικών δαπανών. Ο κίνδυνος εντείνεται από μια σύγκρουση που υπάρχει μεταξύ των επιλέξιμων κριτηρίων και των πραγματικών δαπανών. Και οι δικαιούχοι ε, θα πρέπει να συνυπολογίζουν και το κόστος του προσωπικού και το έμεσο κόστος. Ε, ενώ αυτό δεν συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τον Απρίλιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που έκανε κάποιες προτάσεις για την απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Απλούστευση και διευκρίνηση των κανόνων και των διαδικασιών μπορούν να μειώσουν το περιθώριο σφάλματος και να αυξήσουν τη βεβαιότητα για το σωστό των δαπανών. Και επίσης διευκολύνει τη συμμετοχή των ερευνητών στα προγράμματα και φτάνουμε στους στόχους ε, του ερευνητικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γενική η συνένεση για πολλά θέματα που μπορούν ακόμα να εφαρμόζονται από το γενικό πλαίσιο, το νομικό. Από τις 24 Ιανουαρίου του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα και δράσεις ε, ε, βράχη πρόθεσμα με άμεση αλλά και αναδρομική ισχύ. Ο κύριος Τσουκαλάς, παρακαλώ. Την Επίτροπο για τη λεπτομερή απάντηση. Εξακολουθώ να σημειώνω πάντως ότι με δείγμα 0,4% οι αστοχίες φτάνουν το 4% ή στα 50 δισεκατομμύρια 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελπίζω ότι το μοντέλο δεν είναι γραμμικό και όταν πραγματοποιηθούν έλεγχοι 4% δεν θα βρούμε αστοχίες 40%. Καταλαβαίνω επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο από τη μία μεριά να ζητάμε από την κυρία Επίτροπο να απλοστεύσει τις διαδικασίες διαχείρισης του εβδομού και να προβλέψει απλούστευση για το 8ο, ενώ ταυτοχρόνω ζητούμε λεπτομερέστερους ελέγχους. Αυτό φαίνεται αντιφατικό, όμως νομίζω ότι δεν είναι. Ένα μου φαίνεται καλό, όλοι μας ενδιαφερόμαστε για την έρευνα και ξέρουμε ότι η Ευρώπη μόνο από εκεί μπορεί να σωθεί όπως και τα χώρες μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επιτρόπε, yes, I think our aim has to be that... στόχος μας θα πρέπει να είναι να πλουστεύσουμε όσο το δυνατόν τις διαδικασίες για τους ενδιαφερόμενους, αλλά παρόλα αυτά να εξασφαλίζουμε πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τις λογιστικές ε, διαδικασίες που ακολουθούν έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργήσουν ένα παράλληλο λογιστικό σύστημα, κάτι το οποίο έπρεπε να κάνουν μέχρι σήμερα. Και βέβαια παράλληλα με αυτά ε, καταλαβαίνετε πως δημιουργείται και περιθώριο για και σφάλματα. Όλοι δεχόμαστε πως οι ερευνητές δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα στην κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά ενδιαφέρονται περισσότερο για την έρευνα που οδηγούν στις καταπληκτικές καινοτομίες που βλέπει κανείς όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες το δυνατόν περισσότερο για αυτούς που αφορούν. Ευχαριστώ πολύ να ξεκαθαρίσω σε όσους περιμένουν πως η επόμενη ερώτηση είναι η τελευταία προς την Επίτροπο, γιατί περιμένει και ο Επίτροπος Ποτότσνικ. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι αυτή της κυρίας Τίκαου. Κύριε Μπαλσίτης, ξέρω πως θα την εκπροσωπήσετε. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Κυρία Πρόεδρε, εμείς έχουμε δεσμευτεί να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας, έτσι ώστε ο καρπός τεχνολογίας να φτάσει στην αγορά. Ποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή, όπως το λέμε στην ανακοίνωση για την Ευρώπη, την Ένωση της Καινοτομίας και στην πράξη για τις μικρομεσαίες που εγκρίναμε τον Ιούνιο του 2008, αλλά και στην αναθεώρηση αυτής της πράξης που εγκρίναμε στις 23 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου τρέχοντος. Επίσης, η Πράσινη Βίβλος από τις προκλήσεις της ευκαιρία για το κοινό πρόγραμμα που ενδεχομένως θα ισχύσει στην Ευρώπη για την έρευνα και την τεχνολογία, ορίσαμε τα κομβικά σημεία για το μέλλον της έρευνας και της κοινωνία στην Ευρώπη. Και εδώ θα συμπεριλάβουμε μια σειρά από συγκεκριμένα ερωτήματα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερε ανάγκε των μικρομεσαίων. Ο γενικότερο στόχο του πλαισίου είναι να είναι πρόσβαση εύκολη στα προγράμματα και ελκυστική και κυρίως μιλάω για τις μικρόμεσες επιχειρήσεις. Τι πρέπει να δούμε εδώ. Ε, μία ενιαία θηρίδα εισόδου με κοινή πλατφόρμα υψηλής τεχνολογίας, τυποποιημένους κανόνες, χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα είναι ε, ευθυγραμμισμένα και πιο απλές και συνεκτικές διαδικασίες για την εκταμείευση της χρηματοδότησης. Μετά τις δια βουλεύσεις που έγιναν επί της Πράσινης Βίβλου αποφασίσαμε οι προτάσεις μας να κατατεθούν μέχρι τα τέλη της τρέχουσας χρονιάς. Και έχουμε ήδη στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο εισάγει μία σειρά μέτρων που στοχεύουν συγκεκριμένα σε μικρομεσαίες, δηλαδή ε, δεσμευμένα κονδύλια στον προπολογισμό και τα λοιμά. Και ο προπολογισμό έχει σκοπό να αυξηθεί από το 14,3% σε πάνω από το 15% ως στόχο στον επόμενο προπολογισμό χρειάζονται στήριξη οι μικρομεσαίες και μια καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στο 7ο PP ε, προσφέρεται από τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή για την επιχειρησιακή Ευρώπη ε, και αυτά βέβαια για να διευκολυθούν τα εμπορικά επιμελητήρια, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια και οι αναπτυξιακέ εταιρείε. Έχουμε κατευθυντήρε γραμμέ που έχουν συμφωνηθεί και το δίκτυο αυτό σε συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφή για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο συνδράμουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν, να αυξηθεί το δυναμικό του καλύτερη πρόσβαση προσέλκυση νέων μικρομεσαίων, εταιρικέ σχέσεις, κοινέ δράσεις που είναι ανοιχτές για τις μικρομεσαίες και βέβαια ε, διαβουλεύσεις για τη συμπερίληψη και στόχευση αυτών στα εργασιακά προγράμματα. Αρκετές εκατοντάδες μικρομεσαίες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις για τα προγράμματα αυτά με τη στήριξη τούτου του δικτύου. Σας ευχαριστώ Κύριο Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για τις απαντήσεις σας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν για την ανάπτυξή τους. Ε, υπάρχει συγχρηματοδότηση, αλλά ε, και αυτό ακόμα είναι μεγάλο άχθος για τις επιχειρήσεις αυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια, να εκπονήσει μια απλή σειρά ε, κανόνων έτσι ώστε να μπορούν να ευεργετηθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, γιατί ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί ένα ποσοστό συγκεκριμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τρία συγκεκριμένα μέτρα λέει η απάντηση που δημοσιεύθηκαν τις 24 Ιανουαρίου 2001 που έχουν σαφή επίπτωση στο πρόγραμμα έρευνας By, του προγραμμάτου προγράμματος ε, πλαισίου. Το ένα είναι η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το μισολογικό κόστος ε, και ας πούμε οι υπάλληλοι των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν καταγραφεί οι μισθοί τους μπορούν πλέον να αποζημιωθούν γι' αυτό. Δεύτερον, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούν να αποσαφηνίσουν λύσουν ε, τα σημεία τα οποία δεν είναι αρκετά σαφή και τα οποία δυσκολεύουν τις αιτήσει. Επίσης ε, η δημιουργία μιας πλατφόρμας ε, e-learning που αρχίζει να εφαρμόζεται ήδη από φέτος και που διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική, ε, ε, πραγματικό επιγραμμικό εμπόριο και απελευθέρωση των, ε, του τομέα από συγκεκριμένα προβλήματα και επομένω, ουσιαστικά θα βελτιώσει την θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τη συμμετοχή σας απόψε στην ώρα των ερωτήσεων. Επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση του κυρίου Πόσελτ και απευθύνεται στον Επίτροπο Ποτότσνικ και αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση στις μεγαλοπόλεις της Γερμανίας. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε. Uh, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αξιότιμη κύριε Πόσελτ. Οι αντίστοιχε οδηγίε έχουν ορίσει όρια, ανώτατε τιμέ για ορισμένου ρηπαντέ και με αντίστοιχε προθεσμίε. Πέρα από την προώθηση βέλτιση των πρακτικών, ε, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Εφαρμογής μεταξύ άλλων οργάνων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζεται ε, το, ε, ε, να διεξάγει ελέγχους για το κατά πόσο συμμορφώνονται με τους στόχους τα κράτη-μέλη. Από το 1996 ισχύει η οδηγία και ζητεί από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια γενική στρατηγική με μέτρα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις όταν υπάρχει κίνδυνος ε, υπέρβαση του ορίου των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Ε, και όταν γίνεται αυτή η υπέρβαση, ε, συν το περιθώριο ανοχής, λαμβάνονται μέτρα για να δούμε πώς μπορούν να συμμορφωθούν τα κράτη. Αυτή στιγμή ανακοινώνουν τα προγραμματά τους μέσα σε μία διετία τα κράτη-μέλη από τότε που έχει μετρηθεί η υπέρβαση ή αρμοδιότητα και η ευθύνη ε, για την αντιμετώπιση του θέματος αυτός της ατμοσφαιρικής ρήπανσης είναι στα χέρια των κρατών μελών απολύτως και ε, γράφεται ε, στην επικουρικότητα. Και αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι και οι εθνικές και οι τοπικές αρχές είναι οι πιο ενδεδειγμένες για να αποφασίσουν ποια μέτρα χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την υψηλή ρήπανση της ατμόσφαιρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει λοιπόν τη συμμόρφωση και ε, ακριβώς αυτό, αν ανταποκρίνονται στα όρια, με ποιο τρόπο και ε, πότε. Τα τελευταία στοιχεία που έδωσε η Γερμανία για το 2009 επιβεβαιώνουν ότι 70 από 80 περίπου χώρες, ε, ζώνες που μετράνε την ατμοσφαιρική ρήπανση είναι άνω του ορίου. Οι περισσότερες ζώνες ε, αυτές έχουν μέχρι τις 11 Ιουνίου παράταση φέτος γιατί έχουν προετοιμάσει ένα σχέδιο για την ατμοσφαιρική ρήπαση και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με λεπτομερή μέτρα και ε, προθεσμίες. Το Μόναχο είναι μία από τις ζώνες αυτές, μία από τις πόλεις αυτές. Η παράταση της διορίας ε, δόθηκε με την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές θα προσαρμόσουν το πρόγραμμα ποιότητά τους και θα ε, φέρουν και βραχυπρόθεσμα μέτρα αποτελεσματικά ε, και αν χρειαστεί να ανασταλούν κάποιες δραστηριότητες που επιβαρύνουν ιδιαίτερα την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το διοξίδιο του αζότου, αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζονται και ε, για καταστάσεις πριν από το 2010 με πιθανή παράταση μέχρι το 2014 δεν συνιστούν ε, παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας που ίσχυε τότε, αλλά ε, βοηθούν να δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα τα κράτη-μέλη μέχρι ε, φέτος το Σεπτέμβριο θα πρέπει να υποβάλουν τα σχέδιά τους και τα στοιχεία για το 2010. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πόσελτ. Πολύ καλή, ακριβέστατη απάντηση. Δύο μόνο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί εάν τα κράτη-μέλη πραγματικά εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια και μετρούν με την ίδια αυστηρότητα τις οριακέ τιμές ή υπάρχουν διαφορές. Και δεύτερον, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για τα αστικά κέντρα, πώς μπορεί να περιοριστεί η ατμοσφαιρική ρήπανση. Ευχαριστώ, Επίτροπο. Τα κριτήρια που ισχύουν είναι ίδια για όλες τις χώρες. Όντως βέβαια, λόγω γεωγραφικών συνθήκων, πολλές φορές πόλεις όπως το Μιλάνο στην Ιταλία έχουν ε, μεγαλύτερη δυσκολία να ανταποκριθούν στα κριτήρια αυτά από άλλες χώρες, αλλά είναι ύψη της σημασίας για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίζουμε πως τα επίπεδα υγείας και προστασίας είναι τα ίδια. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το θέμα. Εάν βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα θέματα τοπικά ή περιφερειακά, τότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά και να τα λύσουμε μέσω της συνεργασίας με τις αρχές έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση. Στόχος μας είναι πάντα να βρεθεί μια λύση, δηλαδή να βοηθάμε με αυστηρότητα πάντα. Για τη δεύτερη ερώτηση συνήθως δεν δίνουμε συγκεκριμένες συστάσεις σε καμία από τις πόλεις ή τις περιοχές γιατί πιστεύουμε πως οι αρχές έχουν πολύ μεγαλύτερη γνώση της κατάστασης επιτόπου. Ελέγχουμε εάν ε, έχει επιτευχθεί η συμμόρφωση και συνήθως υπάρχει μια κάπως τυποποιημένη προσέγγιση η οποία φέρνει τα αποθητά αποτελέσματα το οποίο αποτελεί ένα μείγμα διαφόρων μέτρων. Κάποια είναι πιο βραχυπρόθεσμα, άλλα μπορεί να είναι πιο διαστρωτικά. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ερώτηση αυτή της κυρίας Κάπενμπαχ, την οποία αντικαταστά σήμερα ο κύριος Αρσένης. Βιοπικιλότητα και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίτροπε. αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή τελειώνει το πακέτο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι το πλαίσιο για τη στοχευμένη δράση για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της βιοποικιλότητας και νομίζω ότι θα τα καταθέσουμε αρχές Μαΐου. Το σχέδιο στρατηγικής αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εσωτερική διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορώ λοιπόν να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως αποκρίνεται και στην ε, φιλόδοξη εντολή που μας έδωσε πέρσι το Συμβούλιο αλλά και στις παγκόσμιες ε, δεσμεύσεις τις οποίες υπογράψαμε στην Αγκόα πέρσι στην ε, Σύμβαση για την Βιοπικιλότητα. Έχουμε έξι υποστόχους που έχουν ε, ως σκοπό να ε, αντιμετωπίσουν τους βασικούς λόγους της ε, εξαφάνισης βιοποικιλότητας και έχουμε να κάνουμε με συντήρηση, ανανέωση, πράσινες υποδομές, γεωργία, δασοκομεία, αλληλεία, αρπακτικά είδη που εξαπλώνονται και βιοποικιλότητα παγκόσμια. Εάν εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία, η βιοπικιλότητα θα βελτιωθεί και χρειαζόμαστε την κατάλληλη διαχείριση του δικτύου Natura 2000. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς οι μεταρρυθμίσεις στην ΚΑΠ και στην κοινή πολιτική αλίας, όπως επίσης στη μελλοντική πολιτική συνοχή, θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να στηριχθεί η προσπάθεια εξασφάλισης βιοπικιλότητας. Η μεγάλη στόχη του 2020 ζητούν να βοηθήσουμε τα οικοσυστήματα τα οποία καταραίουν και να τα υπηρετήσουμε. Σας εξασφαλίζω λοιπόν πως η στρατηγική αυτή θα συμπεριλαμβάνει δράσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Έχουμε δράσεις λοιπόν για να αυξηθεί η εφαρμογή της ε, οδηγίας για τα οικοσυστήματα και τα πουλιά, όπως επίσης και για την καλή διατήρηση των οικοσυστημάτων των ευρωπαϊκών ειδών. E για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως σκοπό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει μια νέα ανακοίνωση στο θέμα αυτό αργότερα φέτος. Στοχός δεν είναι να υποκαταστήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τις προηγούμενες ανακοινώσεις, αλλά να τις βελτιώσουμε, επικεντρώνοντας στην γενικότερη δομή και γνώση ε, που αποτελούν την υπόθεση εργασίας ε, πάνω στην οποία έχει βασιστεί το κοινοτικό περιβαλλοντολογικό και Και έχουμε διάφορες εναλλακτικέ λύσεις για την ενίσχυση των ελέγχων. Έχουμε και τα εθνικά συστήματα επιθεωρήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως το νομικό πλαίσιο για τις περιβαλλοντολογικές επιθεωρήσεις ήδη βελτιώθηκε τα περασμένα χρόνια, κυρίως μετά την έγκριση της σύστασης για τα ελάχιστα κριτήρια για τις ε, περιβαλλοντολογικές επιθεωρήσεις στα κράτη-μέλη, όπως επίσης και με τη συμπερίληψη κάποιων διατάξεων στην διαστρωτική περιβαλλοντολογική νομοθεσία. Η ανακοίνωση αυτή βρίσκεται ακόμα στα σκαριά και το συγκεκριμένο περιεχόμενο δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα. Θα κάνουμε διαβουλεύσει με του ενδιαφερόμενους βεβαίω και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω τη αρμόδια των αρμοδίων επιτροπών έτσι ώστε τα μέλη να μπορέσουν να εκφράσουν τι απόψει του και να ε, συνεισφέρουν στι δικέ μα προσπάθειε. Σα ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσουμε με τι επιπλέον ερωτήσει. θέλω να σα πω πω όσοι βρίσκονται στην Ολομέλεια ε, να πληροφορθούν πως η επόμενη ερώτηση ε, για τον κύριο Φέρεντς είναι και η τελευταία. Ευχαριστώ πολύ κυρία... Η ερώτηση του κυρίου Χουντή, με συγχωρείτε, είναι η τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαιρόμαστε που βλέπουμε το νέο μανιφέστο και την νέα στρατηγική και βεβαίως ε, το Κοινοβούλιο ε, θα έχει πολλές ε, ιδέες επ' αυτού. Σχετικά με τα θέματα τα οποία συζήτησαμε την Αγκόγια για τη στρατηγική, θα ήθελα να ακούσω τον τρόπο με τον οποίο ε, υλοποιούνται οι ε, αποφάσεις επίσης για το πρωτόκολλο EBS, ε, ποια είναι η πρόοδος, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει στους στόχους να μια ειδική αναφορά πώς προχωρούμε. Επίσης αναφέρατε ότι ε, θα ε, υπέρξουν ε, προσπάθειες για την προστασία της βιοποικιλότητας στα πλαίσια της κοινής βιοικής πολιτικής. Αλλά το Κοινοβούλιο έχει προτείνει συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Επίσης θέλουμε και περισσότερες αναφορές όσον αφορά τις περιοχές 2000. Ναι, και μία επιπλέον ερώτηση από τον κύριο Πόσελτ. Ναι, κύριε Πίτροπε, θέλω να σας ρωτήσω. Σε αυτό το θέμα επικεντρώνεστε πολύ στην προστασία της φύσης και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή ασχολείστε και με όλα τα κατοικίδια, ζώα, τα οικόσιτα και τα διάφορα άλλα φυτά, όχι τα άγρια, τα ήμερα που επίσης απειλούνται πάρα πολύ. Και άλλη συμπληρωματική ερώτηση. Well, um, thank um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι. Μιλάμε για βιοπικιλότητα. Ένα από τα ζητήματα τα οποία είναι επίγοντα αυτή τη στιγμή μεταξύ πολλών κρατών μελών, το των οποίων και το δικό μου, είναι ότι έχουμε χαμηλότερους στόχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προστασία της φύσης και την νομοθεσία αυτή. Θα ήθελα να μου πει ο Επίτροπος εάν συμφωνεί ότι μπορούμε να φτάσουμε σε χαμηλότερους στόχους ή αν πρέπει να μείνουμε στους παρόντες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Επίτροπος παρακαλώ. Ευχαριστώ και τους τρεις ε, παρεμβαίνοντες. Όσον αφορά την ε, Ναγκόγια, ε, όσον αφορά το EBS προχωρούν καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε πρόβλημα εκεί. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα με τη μετάφραση, αλλά όσον αφορά την ουσία δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι καλή τροχιά. Και προτιθέμεθα να ξεκινήσουμε την προετοιμασία της ε, ε, νομοθεσία ε, μετά την ε, διαδικασία επικύρωση, Υπάρχουν πολύ λίγα εμπόδια, τα ξεπερνάμε. Όσον αφορά τι προστατευμένε θαλάσσιε περιοχέ, όντω είναι γεγονό ότι έχουμε μείνει πίσω. Προσπαθούμε να πιέσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά είναι προφανέ ότι και λόγω των δεσμεύσεων τη ε, Ναγκόγια πρέπει να γίνουν περισσότερα στην Ευρώπη όσον αφορά την παρούσα κατάσταση και βεβαίω και λόγω του, της ίδιας της Natura 2000. Ε, κοινή πολιτική και Natura 2000. Προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο έτσι ώστε ε, να μπουν και στο πρώτο και στο τρίτο πυλώνα με τον σωστό τρόπο να αντιμετωπιστούν ε, και ότι εν πάση περιπτώσει στην μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική θα υπογραμμιστούν τα ζητήματα αυτά και θα υπάρξει ιδέουσα προσοχή και ο Επίτροπος Χέντεγκαρτ και εγώ ίδιος ε, έχουμε ε, αναφερθεί στα προβλήματα αυτά σε μια επιστολή την οποία σας έχουμε αποστείλει. Ε, για την ερώτηση του κυρίου Πόσελτ μπορώ να πω το εξής η προστασία βάσει της Natura 2000 έτσι όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή ε, προστατεύει 18% περίπου ε, της, του ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτά είναι τα Natura 2000 και μετά έχουμε και δύο οδηγίες, μία για, τους, για τα πουλιά και μία για τα οικοσυστήματα όπου σαφέστερα αποσαφηνίζονται τι προστατεύεται ε, και σε ποιο επίπεδο προστασίας. Στην ουσία πρόκειται για ευρία ε, νομική βάση που δεν ασχολείται έτσι πολύ εξειδικευμένα με συγκεκριμένα είδη. Θέλαμε ευρεία προστασία και είναι γεγονός βέβαια ότι πολλά είδη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν διαπιστωθεί ε, ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Όσον αφορά την ερώτηση για τους στόχους, η απάντηση είναι νομίζω απλή. Αυτή τη στιγμή δεν εστιάζουμε στην μείωση των στόχων αλλά σε καλύτερη αντιμετώπιση των στόχων Natura 2000 και ε, θέλουμε να ε, υπάρχει αρκετή ε, χρηματοδότηση σε αποθεματικό έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση. Του κυρίου Χουντή και αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Αξιότιμοι βουλευτέ, αγαπητέ κύριε Χοντή, η νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα έχει μια ιεραρχία πέντε βαθμίδων για τη διαχείριση. Η πρόληψη των απορριμμάτων είναι η πιο επιθυμητή λύση. Μετά η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση και άλλοι τρόποι ανάκτησης και σε ενεργειακό επίπεδο με ε, τελευταία έσχατη λύση πραγματικά τη χωματερή, την υγειονομική ταφή. Υπάρχει δυνατότητα ε, απόκλησης από την ιεραρχία, αλλά τα κράτη θα πρέπει να δίνουν βάσιμη αιτιολόγηση. Άρα, η γενομική ταφή ε, που είναι η έσχατη λύση θα πρέπει να θεωρείται από το κράτος μέλος ακριβώς ε, η λιγότερο επιθυμητή. Το χαρτί και το γυαλί είναι υψηλής ποιότητας υλικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ε, δευτερογενείς ε, πρώτες ύλες ε, από τη βιομηχανία. Γι' αυτό θα πρέπει στην πηγή να γίνεται η διαλογή και αυτή είναι η πιο επιθυμητή μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων. Με βάση την οδηγία πλαίσιο, τα κράτη-μέλη μέχρι το 2015 θα πρέπει να συλλέγουν χωριστά το πλαστικό, το μέταλλο, το γυαλί και το χαρτί. Βεβαίως υπάρχει κάποια ευελιξία, κάποιο περιθώριο ε, στην αποκομιδή ε, αναχώρα με βάση κάποιες ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ε, δεν υπάρχουν ε, τεχνολογίες υψηλής ποιότητας και πιο σύγχρονες. Πάντως η πιο φτηνή και πιο εύκολη μέθοδος είναι η διαλογή στην πηγή για να ε, διαχωρίζονται τα υλικά και οι πρώτες ύλες από τα απορρίμματα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις παράνομες χωματερές και όπως γνωρίζετε το 2015 ε, τα δικάστηκε από το ΔΕΚ για το τεράστιο αριθμό ε, χωματερών που λειτουργούν παράνομα στη χώρα. Δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα, ωστόσο το Δεκέμβριο του 2010 οι ελληνικές αρχές έδωσαν πρόγραμμα δράσης με βάση το οποίο όλες οι παράνομες χωματερές θα κλείσουν μέχρι το ε, τέλος Ιουνίου 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει αυτό το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων ε, χώρων υγειονομική ταφή υπό τον όρο ότι είναι έσχατη ε, λύση, αναπόφευτη λύση. Ε, στο βαθμό βέβαια που τηρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές για την ταφή των απορριμμάτων. Βάσει την αντίστοιχη οδηγία. Αυτό ήδη από μόνο του συνιστά πρόοδο σε σύγκριση με την ε, ε πρακτική παράνομης χωματερής. Ε, ε, ε εμείς αθαρρύνουμε την ελληνική κυβέρνηση για την κατασκευή των χιτά και των χιτή που συγχρηματοδοτούνται, αλλά θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει και πέρα από αυτή την επιλογή διαχείρισης αποβλήτων να ξεφύγει από τα χιτά και χιτή και να φτάσει σε πιο σύγχρονες μεθόδους που βασίζονται στην ανάκτηση και την ανακύκλωση. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες στατιστικές της Eurostat στην Ελλάδα, περίπου 82% ε, των ε, δημοτικών, των αστικών αποβλήτων καταλήγουν σε χωματερές, ενώ στο μέσο όρο της Ένωσης είναι 38%. Επιπλέον, η ανακύκλωση στην Ελλάδα έχει πολύ χαμηλές επιδόσεις. Μόλις 17% των αστικών αποπλήτων ανακυκλώνονται. Είναι ύψιστη προτεραιότητα η εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για μένα προσωπικά. Θα ε, παρακολουθούμε τα κράτη-μέλη στα προγράμματα, στα σχέδιά τους και τη διαχείριση. Περιμένουμε ένα ενημερημένο πρόγραμμα από την Ελλάδα και επιπλέον παρακολουθούμε πολύ στενά ε, το πρόγραμμα δράσης και τη διαδικασία ε, ε, κλεισίματος όλων των παράνομων χωματερών και εκείνων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα έργα που χρηματοδοτούμε συνάδουν με τους στόχους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία μας για τα απόβλητα. Στην περίπτωση της Ελλάδας είναι απαραίτητο να μειωθεί η υγειονομική ταφή ε, και να αυξηθεί η ανακύκλωση με χωριστή αποκομιδή και διαλογή στην πηγή. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία γιατί μπορεί να δημιουργήσει και θέσεις απασχόλησης και ε, σε όλη τη χώρα. Επίσης θα πρέπει να ε, διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές και τέλος θα ήθελα να πω στον αξιότιμο βουλευτή ότι αύριο ε, θα πάω στην Ελλάδα και σε δύο μέρες θα έχω πλήρη εκτενή επίσκεψη και θα συζητήσω όλα τα θέματα σε βάθος με τους ε, ε, αρμοδίους. Ο κύριος Χουντής, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η τελευταία αναφορά του Επιτρόπου μου δίνει κάποιες ελπίδες. Αφού λοιπόν κύριε Επίτροπε θα πάτε αύριο στην Ελλάδα, επισκεφτείτε μια περιοχή κοντά στην Αθήνα, όπου για τέσσερις μήνες τώρα υπάρχει καθημερινή σύγκρουση των κατοίκων με αστυνομικέ δυνάμει που στρατοπεδεύουν εκεί με τραυματισμού και άλλο σχετικά με τη διενέργεια την εγκατάσταση χιτά χιτή έτσι όπω τα αναλύσατε και με το ότι πρέπει να κλείσουμε τι χωματερέ. η ερώτηση είναι εφόσον είναι η χειρότερη από τι αποδεκτέ λύσει γιατί κάνετε δεκτέ ε, μελέτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου σε πολλέ περιπτώσει και σε αυτή που ενδεχομένω επισκεφτείτε έχουμε ουσιαστικά απορρίμματα που καταλήγουν σε ρέματα. αυτό είναι σκάνδαλο και η καταστροφή που γίνεται για το περιβάλλον αν δεν παρέμβετε αν δεν σταματήσετε αυτό το οικονομικό σκάνδαλο διότι συγχρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή ένωση δεν θα λυθεί το πρόβλημα. σας παρακαλώ παρεμβείτε πιο άμεσα διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο θεωρητικά όπως τα αναλύσατε και σας ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ έχετε μία επιπλέον πρόσκληση που σας απευθύνεται κύριε Επίτροπε. Ναι, θα πάω, θα πάω. Είναι κοντά στην Αθήνα και την πρώτη μέρα θα κάνω και μία συζήτηση με τρεις επιτροπές του Ελληνικού, της Ελληνικής Βουλής, όπου σίγουρα θα συζητήσουμε και το θέμα αυτό. Το γνωρίζω. Και επίσης ξέρω και ποια είναι η σοβαρότητα του θέματος. Να σας πω λοιπόν πως και να σας εξηγήσω γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε υπέρ αυτής και μάλιστα προχωράμε και σε συγχρηματοδότηση παρόλο που θεωρούμε πως από τις επιλεγόμενες εναλλακτικές λύσεις θα έπρεπε να είναι η λιγότερο προτιμητέα. Πρώτα απ' όλα, το βασικότερο το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι λοιπόν πως με κάθε τρόπο εξασφαλίζονται. Και είναι σημαντικό να βρούμε την καλύτερη δυνατόν εναλλακτική λύση. Γιατί καμιά φορά είναι απαραίτητο κανείς να προχωρήσει σταδιακά, βήμα-βήμα. Από τα στοιχεία τα οποία λαμβάνω από όλη την Ευρώπη, βλέπω πως όταν μία χώρα ξεκινάει μία σοβαρή προσπάθεια διαλογής ε, και διαχωρισμού υλικών, τότε γρήγορα επιτυχαίνει ένα γρήγορο ρυθμό ανακύκλωσης ε, και ε, μειώνεται πολύ γοργά η υγειονομική ταφή. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αυτή την ε, ξεχωριστή, το διαχωρισμό στην αποκομιδή. Γιατί καταλαβαίνω πως αυτή τη στιγμή η μοναδική λύση είναι η οικονομική ταφή. Και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να το δεχτούμε και πρέπει άρα να προσφέρουμε και χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τη συμμετοχή σας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για ερωτήσεις. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις απαντηθούν γραπτά. Λίγοι λοιπόν το τμήμα αυτό της συνάντησης. Ευχαριστώ. Και διακόπτεται η σύνδεση μέχρι τις 9.